Αγαπητοί συνάδελφοι, άρχεται η συνεδρίαση. Θα ήθελα να σας πω ότι ο πρόεδρος Αλμπερτίνη δυστυχώς κολλείεται σήμερα παρευρεθεί και ζητεί συγγνώμη γι' αυτό. Ε, σας υποβάλλω την ημερήσια διάταξη, τη γνωρίζετε. Σήμερα το πρωί θα εξετάσουμε πρώτα την πρόταση ψηφίσματος για την Ισλανδία είναι για δεύτερη φορά συζήτηση. Στόχος συζήτησης είναι η εξέταση των τροπολογιών, 20 περίπου τροπολογίες κατατέθηκαν, ξέρω με τους συναδέλφων για την έκθεση αυτή, του κυρίου Κριστιαν Πρέντα. Πού είστε κύριε Πρέντα? Ορίστε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω ρουμανικά. Κάναμε μια πρώτη συζήτηση στην Επίτροπή μας στις 10 Φεβρουαρίου. Έκτοτε έχουν συμβεί δύο σημαντικά γεγονότα σχετικά με την Ισλανδία. Πρώτον, η συμφωνία ISAVE ε θα υποβληθεί σε δημοψήφισμα στις 9 Απριλίου, έτσι αποφάσισε ο πρόεδρος της χώρας. Και λαμβάνοντας υπόψη ε, αυτή την κατάσταση υπέβαλα στη συνέχεια προφορική τροπολογία στην παράγραφο 10 του κειμένου που είχαμε συζητήσει το Φεβρουάριο και θα σας την αναγνώσω. Η Ισλανδική Βουλή με μεγάλη πλειοψηφία στις 17 Φεβρουαρίου 2011 ε, λαμβάνει υπόψη την ε, απόφαση του Προέδρου της χώρας ε, να ε, υποβληθεί σε δημοψήφισμα η πρόταση αυτή για να τερματιστεί η διαδικασία προσβολής, η παραβιάση που ξεκίνησε στις 26 Μαΐου του 2010 από την ΕΖΕΣ. Τελειώνει η παράθεση και νομίζω ότι είναι σημαντικό να προσθέσουμε εδώ ότι η Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Ισλανδών είναι υπέρ της νέας αυτής συμφωνίας. Ε, οπότε και θα υπερψηφίσουν φαντάζομαι στις 9 Απριλίου. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι απέτυχε ο έβδομος γύρος διαπραγματεύσεων να βάγισε Ευρωπαϊκή Ένωση, Νορβηγία, Ισλανδία και Νήσι Φερόε για ε, την κοινή διαχείριση των αποθεμάτων ε, σκόμβρου. Ε, ε, σας παραθέτω και πάλι την αντιστοιχή παράγραφο. θα ρίνουμε την Ισλανδία να διατηρήσει το ταχύ βηματισμό της ε, στις διαπραγματεύσεις με στόχο να έχουμε μια ποσόστοση βιώσιμη στο μέλλον και αηφόρο και ε, αυτή είναι η τροπολογία που έχω καταθέσει προφορική για αυτό το δεύτερο στοιχείο. Υποστηρίζω ε, τις περισσότερες τροπολογίες των συναδέλφων, διότι ε, συμπεριλαμβάνουν πολλά χρήσιμα στοιχεία και τα δέχομαι. Υπάρχουν όμως και τροπολογίες οι οποίες δεν μπορώ να δεχτώ. Παράδειγμα, η παριθμόν 1 Τάρατ και ε, Σαρζεντίνη. Νομίζω ότι αυτή η πρωτοβουλία δεν συνδέεται άμεσα με τις ε, ε, διαπραγματεύσεις προσχώρησης και το δεύτερο τμήμα κάνει αναφορά στην εσωτερική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πάλι δεν θεωρώ ότι έχει καμία σχέση αυτό με το ψήφισμα. Στην τροπολογία παριθμών 2 που έχει υποβάλει ο κύριος Δέβα, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας λόγος να φοβούμαστε ε, ότι ε, θα επιταχυθούν οι διαπραγματεύσεις γιατί έρευνα για την iSave. Είχε αρκετό χρόνο στη διάθεσή της Ερευνητική Επιτροπή η ε, έκθεση που προέκυψε για την κρίση και τη χρηματοπιστωτική και τη τραπεζική που συγκλώνησε τη χώρα το 2008. Ε, είναι αρκετά εμπεριστατωμένη και εκτενής. Έχει μελετηθεί πολύ. Επίση πρέπει να σας πω ότι τώρα η ανάκριση και η έρευνα που γίνεται ε, κατά του πρώην Πρωθυπουργού προχωράει με κανονικούς ρυθμούς. Σε ό,τι αφορά τώρα την τροπολογία υπαριθμών 10 ασχολείται με το θέμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλίας. Νομίζω είναι πάρα πολύ πρόημο το στάδιο να συζητήσουμε αυτό το θέμα, γιατί είμαστε στη διαδικασία ελέγχου ακόμα, screening, screening συγγνώμη, και δεν έχουν αρχίσει οι διαπραγματεύσεις και δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε την ιδέα αυτή τη στιγμή να εξαιρεθεί, να αποκλειστεί η Ισλανδία από ε, αυτό το σκέλος του κοινοτικού και εκτιμένου. Και τέλος, ε, απορρίπτω διάφορες τροπολογίες που ζητούν πλήρη ή μερική απάλληψη ε, της αναφοράς της κοινή γνώμης στην Ισλανδία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το θέμα της ένταξης της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορώ να δεχτώ τέτοιες ε, τροπολογίες, γιατί ό,τι έχει να κάνει με την κατάσταση της κοινή γνώμης είναι σημαντικό. Νομίζω δεν ασφαλώ όταν λέγω ότι η κοινή γνώμη είναι πάρα πολύ σημαντική πολιτική πτυχή όταν ζητούμε, συζητούμε για την πρόσβαση της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν άποψη για αυτό το θέμα Ιδιαίτερα σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωβαρομέτρου προέκυψε ότι 56% των Ισλανδών ε, εμπιστεύονται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενώ μόλις 28% εμπιστεύονται τη δική τους Βουλή. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Watson. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την έκθεση που μας παρουσιάζει. Ε, νομίζω πιο μακριά από την Ισλανδία δεν θα μπορούσε να ήταν η γενέτειρα του εισηγητή. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεται το μέγεθος των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα οι φιλελεύθεροι δεν έχουν καμιά σοβαρή ένσταση για το περιεχόμενο της έκθεσης. Θα υποβάλουμε μια-δύο τροπολογίες για τη διατύπωση. Αλλά καταρχήν υποστηρίζουμε το σχέδιο. Τρία είναι τα βασικά ζητήματα κατά τη γνώμη μας. Πρώτον, η βούληση του λαού του ίδιου της Ισλανδίας να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση Περιμένουμε την επίσημη έκφανση, απόδειξη της βούλησης αυτής. Δεύτερον, αποζημίωση από τις τράπεζες. Είναι καλή η συμφωνία στην οποία κατέληξαν τα εμπλεκόμενα μέρη κατά τη γνώμη μας και ομολογουμένως κάποιοι από τις τοπικές αρχές και όσοι διερεύνησαν τις Ισλανδικές τράπεζες ε, θα ήταν ε, προτιμότερο να είχαν μεριμνήσει περισσότερο όταν έκαναν τις επενδύσεις τους και να μην ασχολούνται μόνο με τις ε, αποδόσεις ε, των ε, επενδύσεων. Και όπως είπε και ο εισηγητής, βέβαια υπάρχει μία λεπτομερής έκθεση γι' αυτό και εν γέννη μας ικανοποιεί. Τρίτο θέμα, Αλία φαλαινοθυρία συγκεκριμένα. Θα πρέπει να εξετάσουμε αυτό το θέμα κατά τη διάρκεια και τη συνέχεια των διαπραγματεύσεων. Θα πρέπει να δείξουμε ευαισθησία, ε, διότι είναι μια πατροπαράδοτη Ισλανδική βιομηχανία. Αυτόχρονα βέβαια θα πρέπει να ε, συμμορφωθούμε με τις απαιτήσει ε, που έχουμε προβλέψει για την ε, περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Μία ερώτηση για την παράγραφο 6 θα ήθελα να θέσω στον εισηγητή σχετικά με τα πολιτικά κριτήρια σχετικά με το ρόλο του Υπουργού Δικαιοσύνης για τους διορισμούς δικαστικών αξιωματούχων. Είναι σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, να αντιληφθούμε ποια είναι η φύση αυτής της μικρής χώρας της Ισλανδίας. Όλοι γνωρίζουν τους πάντες στην Ισλανδία και τελικά κάποιος πρέπει να φέρει την πολιτική ευθύνη για τις αποφάσεις ε, που λαμβάνονται. Και γι' αυτό ε, το λόγο, αυτό το σύστημα βάσει του οποίου ε, προσδίδεται ιδιαίτερη ευθύνη στον Υπουργό Δικαιοσύνη ανεπτύχθη υπέρμετρα και πρέπει να το συζητήσουμε αυτό με τους Ισλανδούς και να δούμε αν μετά τη συζήτηση θα προτίθενται να τροποποιήσουν το σύστημα. Όμως αναγνωρίζοντα την ιδιάζουσα ε, φύση αυτής της μικρής κοινότητας, τη μικρής ε, χώρας, ε, θα πρέπει να δείξουμε κατανόηση για αυτά τα χαρακτηριστικά της Ισλανδίας. Ευχαριστούμε κύριε Βότσον, η κυρία Χάουταλα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω να ρωτήσω αν ε, θα μπορούσε ο εισηγητή και λοιπέ πολιτικέ ομάδε να εξετάσουν ε, με προσοχή και ευμενώ στην τροπολογία ένα των Πρασίνων, βάσει τη οποία ε, υποστηρίζεται η πρωτοβουλία για τα μέσα μαζική ενημέρωση, πρωτοβουλία τη Ισλανδική κυβέρνηση. Έχουν γίνει πολύ ενδιαφέροντα πειράματα και νομικό πώ στην Ισλανδία για να βρεθεί ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και την ελεύθερη πρόσβαση στι πληροφορίε των ΜΜΕ. Θα μπορούσατε να εξετάσετε λοιπόν αυτή η τροπολογία, ίσως να καταλήξουμε σε μια προφορική, αλλά να διατηρηθεί η ουσία παρακαλώ, ε, η δυνατόν στην τελική έκθεση. Σας ευχαριστούμε κυρία μου. Δεν βλέπω να υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις. Ο κύριος Φέρν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συγχαρητήρια προ τον εισηγητή. Είναι εξαιρετική η έκθεση. Είμαι πραγματικό μέλο τη Επιτροπή. Εγώ είμαι στην Επιτροπή Προπολογισμών και μόνιμο εισηγητή για τη διεύρυνση και γι' αυτό με ενδιαφέρει το ζήτημα. Βασικά πιστεύω πω οι προτάσει σχετικά με το πώ θα χειριστούμε τι τροπολογίε δεν μα δημιουργούν πρόβλημα. Θα ήθελα άλλο ιδιαίτερο να τονίσω την ε, σημασία μια ενδεχόμενη ε, απόρρεψη τροπολογία 17 για τα μέσα μαζική ενημέρωση. Νομίζω ότι θα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα η τροπολογία για το όλο θέμα. Θα επανέλθω. Ε, το Μάιο θα στείλουμε αντιπροσωπή από την Επιτροπή μα. Δεν μπορέσαμε να συντονιστούμε με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Δεν πειράζει γιατί δεν μπορούμε να πάμε το φθινόπωρο. Έχουμε διαπραγματεύσει για τον προπολογισμό. Άρα πρέπει να πάμε το Μάιο. Το σημαντικό είναι να πούμε ότι από πλευρά τη Ισλανδία υπάρχει βούληση να βρουν λύσει για τα βασικά του προβλήματα. Είμαι πεπισμένη γι' αυτό για τα οικονομικά ζητήματα. Είναι πολύ σύνθετα και θα κρίνουμε από την έκβαση και του δημοψηφίσματο πώ θα κινηθούμε. Όμω θα πρέπει να καταδείξουν ότι επιθυμούν να βρεθεί μια λύση για δύσκολα ζητήματα όπω τα αλλιευτικά. Δεν ζητούν ε, βαρεκλήσει, δεν ζητούν ξεχωριστέ ε, ε, μεμονωμένε λύσει. Θέλουν να διαπραγματευτούν. Πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης μπορεί να είναι μεγάλα του για την Ευρώπη η Ισλανδία. Πέρα από τη στρατηγική σημασία είναι πολύ προηγμένη η κοινωνία τους με αυξημένε γνώσεις για σημαντικά θέματα όπως διαχείριση του θαλασσίου, βίου, ενέργεια, ε, ε, αλία κτλ. Εμείς μπορούμε να μάθουμε από αυτούς για αυτά τα ζητήματα. Όμως, όμως και το είπε και ο κ. Γότσον και άλλοι, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μοναδική περίπτωση η Ισλανδία, πολύ προηγμένη, πολύ σύγχρονη κοινωνία. Ταυτόχρονα όμως αυτή η κοινωνία ε, ε υπερασπίζεται τη γλώσσα, την κουλτούρα της, τον τρόπο ζωής της, ε, με τα και άρα εμείς πρέπει να βρούμε ευέλικτες λύσεις. Και υπάρχουν και δύο τομείς που δεν προαναφέρθηκαν, που όμως θα δημιουργήσουν θέματα. Η γεωργία και η περιφερειακή ανάπτυξη, ανάπτυξη υπάρχουν ναι, επαρχίε στην Ισλανδία που διαφέρουν πάρα πολύ από την κατάσταση που βλέπουμε στο Ρέικιαβεκ, παραδείγματο χάρη. Άρα θα πρέπει να είμαστε διαλλακτικοί, να βρούμε λύσει και για αυτά τα προβλήματα και γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε ενημέρωση. Και άρα είναι σοφό να απορριφθεί αυτή η τροπολογία 17 κατά τη γνώμη μα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Αν δεν θέλει κανένα άλλο συνάδελφο το λόγο, ο εισηγητή μα για να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους. Πάρα πολύ σύντομα μου επιτρέπετε. Σε ό,τι αφορά την παράγραφο 6 που ανέφερε ο κύριος Γότσον, η παράγραφος αυτή είναι θετική. Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για τις προσπάθειες που καταβάλουν οι Ισλανδοί για την ε, ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Το θέμα των διορισμών ε, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι κάτι που ρώτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε αυτό. Γι' αυτό ψηφίσαμε στην παράγραφο αυτή και σημειώνουμε, μάλλον σημειώνουμε τις προόδους που κάνουν οι Ισλανδικές αρχές ε, διατηρώντας πάντα τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της πάρα πολύ μικρής κοινότητας που ε, είναι αυτό το κράτος τώρα. Σε σχέση με τα όσα είπε η κυρία Χάουταλα, την πρώτη τροπολογία. Όπως σας είπα προηγουμένως, φρονώ ότι αυτή η πρωτοβουλία για τα μέσα ενημέρωσης δεν είναι κάτι που έχει να κάνει με τη διαπραγμάτευση. Και για το δεύτερο, μάλλον το τελευταίο τμήμα της τροπολογίας του κυρίου Τάραντ και της κυρίας Αρχεντίνη προτείνει να αλλάξει το κεκτημένο ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι γίνεται αυτό, πώς θα το κάνουμε. Ε, κατά τα λοιπά θα μπορούσαμε να δούμε αν με άλλο τρόπο μπορούμε να δεχτούμε την τροπολογία. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον κύριο Φέρμ για τα σχόλιά του. Τώρα σε ό,τι αφορά την τροπολογία 17 που ανέφερε και εκείνος, Κατά την άποψή μου δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό, να το διαγράψουμε και να απαλληφθεί αυτό που αναφέρει παράγραφος 31. Δεν μπορώ να δεχτώ καθόλου την τροπολογία 17. Ευχαριστώ πολύ. Διαφωνούμε από ό,τι φαίνεται. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Σας ενημερώνω για την ψηφοφορία. Θα γίνει το απόγευμα αφού τελειώσει η ανταλλαγή απόψε με την κυρία Άστον. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Πρώτη συζήτηση για την έκθεση πρωτοβουλίας της κυρίας ε, Μουνής. Ο, κόσμος, ε, ο Παγκόσμιος Φορέας και πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει στις πολυμερείς οργανώσεις μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας. για να βοηθήσουμε την εισηγήτρια να κάνει τις προτάσεις, αναθέσαμε εξωτερική μελέτη. Και πριν δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, θα ήθελα να καλωσορίσω τους δύο εμπειρογνώμονες μας που έκαναν τη μελέτη αυτή, η οποία διανέμεται στην αίθουσα. Ο κύριος Μανουέλ Ντελαρόκα και Βινθέντε Παλάσιο από το ε, Ισπανικό Ίδρυμα Αλτερνατίβα, εναλλακτικέ ε, λύσει. Εναλλακτικέ προτάσει. Παρακαλώ σύντομα να μα παρουσιάζετε τα αποτελέσματα τη έρευνα αυτή. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μας καλέσατε να παρουσιάσουμε την έκθεση αυτή, τη μελέτη για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις πολυμερείς οργανώσεις, θα πρέπει να εντοπίσουμε τα προβλήματα, τις ευκαιρίες και να διερευνήσουμε και το πεδίο δράσης. Η έκθεση αυτή δεν είναι ολοκληρωμένη, δεν είναι πλήρης. Πάντα είμαστε πρόθυμοι να ακούσουμε ερωτήσεις και υποδείξεις από πλευρά σας και προτάσεις. Βασικό στόχος της έκθεσης αυτής ήταν να διερευνήσουμε τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μεγιστοποιήσει τον ρόλο της σε πολυμερείς οργανώσεις μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Για το λόγο αυτό επικεντρωθήκαμε πρώτα στη νομική βάση της συνθήκης της Λισαβόνας μέσω μελέτης των νέων αρμοδιοτήτων ε, της Ένωσης στα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης. Προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε τη στιγμή και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αλλάζει. Αυτό σημαίνει να αποτυπώσουμε τη δυναμική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς θα είναι μεγαλύτερη προβολή της, μεγαλύτερη ισχύ της ε, διεθνώς. Επιλέξαμε λοιπόν κάποιες βασικές πολυμερείς οργανώσεις οργανισμούς, το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, το G20, το ΝΑΤΟ και τον ΟΑΣΕ που είναι κυρίως οργανισμοί ασφαλείας. Δεν έχουμε ε, την αξίωση να καλύψουμε σε 25 σελίδες όλες τις ε, πολυμερείς διεθνείς οργανώσεις. Επίσης προσπαθήσαμε να ε, προβληματιστούμε για το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στις δυνατότητες και τις πραγματικές δράσεις στην κοινή εξωτερική δράση. Η βασική θέση και η βασική παραδοχή είναι ότι η πολυμερή συνεργασία δεν ε, πηγαίνει καλά, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αξιοποιεί πλήρως το δυναμικό της διεθνώς και θα πρέπει η διαδικασία αυτή να θεωρείται ως ε, διαδραστική ε, προσπάθεια, συνεργασία των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων αφενός και αφετέρου τον εσωτερικό συντονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για βασικές θέσεις για ενίσχυση του μηχανισμού συντονισμού γιατί υπάρχει αυτή η διαμάχη μεταξύ των δαρβενιστών και των λεγόμενων λειτουργιστών και θα πρέπει και οι δύο πλευρές να εργάζονται ε, σωστά. Η εξωτερική ε, αντιπροσώπευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, γνωρίζει μια παράδοξη κατάσταση. Από τη Λισαβόνα και μετά έχει μειωθεί η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντί να αυξηθεί. Υπάρχουν και προβλήματα και προσκόμματα που ε, προβάλλουν κάποιες χώρες ε, μέλη και αυτό καταλήγει σε κοινό εκπροσώπηση στις διεθνείς αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναβαθμίσει το σημερινό της καθεστώς σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς. Ε, αν είναι ε, να γίνει πλήρες μέλος, ας πούμε, ή η συμμετοχή της. Και η Αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρία Άστο, θα πρέπει να αξιοποιήσει τη θέση τη αυτή για να αναβαθμίσει το ρόλο και την παρουσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση με συνεκτικέ πολιτικέ εξωτερική δράση, ανθρωπιστική συνεργασία, για παράδειγμα, ε, η αναπτυξιακή εμπόριο, μαζί με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Και επίσης η βελτίωση τη υπηρεσία εξωτερικής δράσης ως προς το προσωπικό τη δεν θα πρέπει να είναι ποσοτική αλλά ποιοτική. Όχι περισσότερους υπαλλήλου, αλλά ενίσχυση ε, για να ε, είναι ταχύτερη η εκπροσώπηση και η αντίδραση ε, στους διεθνείς οργανισμούς όπως είναι τα Ηνωμένα Έθνη ή χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που είναι αργή η δράση μας. Έχουμε και προτάσεις για το Κοινοβούλιο. Παράδειγμα. Χρειαζόμαστε κοινό μηχανισμό συμφωνίας, ένα πρωτόκολλο δράσης, όπως δείχνει η σημερινή κρίση στη Λιβύη και πιστεύουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να ε, δίνει τακτικά συστάσεις μέσω εκθέσεων στην ε, ύπατη εκπρόσωπο. Για τα οικονομικά θα τα πει ο συνάδελφος Ρόκα, αλλά αυτό που χρειάζεται είναι απόλυτη προτεραιότητα να μεταρρυθμιστεί το σύστημα για το Ηνωμένα Έθνη. Ε, για τη Γενική Συνέλευση θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει ένα προηγμένο καθεστώς ε, παρατηρητή. Ήδη γίνονται κινήσεις από το περασμένο Σεπτέμβριο και ε, να ενισχύσουμε τις δυνατότητες των λεγόμενων περιφερειακών οργανισμών, περιφερειακής ολοκλήρωσης. να ξεφύγουμε δηλαδή από την εθνοκεντρική λογική που έχει ο Οργανισμός Εθνών, να περάσουμε σε περιφερειακή διάσταση. Δεν ζητάμε μία έδρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, βράχει πρόθεσμα, αυτό δεν θα ήταν ρεαλιστικός στόχος, αλλά ζητούμε ε, ε, αύξηση των μονίμων μελών στο Συμβούλιο Ασφαλείας, να υπάρχει υπερενισχυμένη πλειοψηφία για να καταργηθεί το βέτο και να προχωρήσουμε περισσότερο ένα βήμα ε, προς την Ευρώπη της άμυνας, πράγμα που είναι απαραίτητο για την παγκόσμια ασφάλεια. Ε, Πρόεδρε, ευχαριστούμε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συγκεκριμένα την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ε, για την πρόσκληση, ούτως ώστε να παρουσιάσουμε τον προβληματισμό, τι σκέψει μας και τα αποτελέσματά μας σχετικά με το ρόλο στη διεθνή σκηνή της Ευρωπαϊκής Ένωση. Θα ήθελα, εν συντομία, να σχολιάσω τις συστάσεις μας ε, για τις τρεις οργανώσεις που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Παγκόσμια Τράπεζα και η Σύνθεση G20. Για το ΔΝΤΑΦ, το Θεωρούμε ότι υπάρχει μεγάλη ασυνέχεια, διότι έχουμε ένα υπερεθνικό σώμα με παγκόσμια συμφέροντα, ενώ ε, τα μέλη είναι εθνικές οργανώσεις ε, υπάρχει αποκλειστική αρμοδιότητα για την ε, Παγκόσμια Τράπεζα για θέματα όπως ε, η μακροφορολογική πολιτική είναι θέματα μεικτής αρμοδιότητας, αλλά υπάρχει συντονισμός. Ε, πάντως ε, δεν υπάρχει καμία εκπροσώπηση της Ένωσης ούτε με το καθεστώς παρατηρητή. Λοιπόν, για την νομισματική πολιτική στη ζώνη ευρώ δεν υπάρχει φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Παγκόσμια Τράπεζα διότι δεν εκπροσωπείται στο εκτελεστικό συμβούλιο ούτε του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ούτε της Παγκοσμίας Τράπεζας και για τα υπόλοιπα θέματα στερείται επίσημη εκπροσώπηση Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε το θέμα του Διοικητικού Συμβουλίου τη Παγκόσμια Τράπεζα, αν βασιστούμε σε εκλογικέ περιφέρειες για τι ψήφου των μικρών χωρών, είναι μία λύση. Δηλαδή, οι πέντε βασικοί μέτοχοι έχουν ε, μεμονωμένε έδρε. Ε, με την εξαίρεση τη Γερμανία, τη Γαλλία και του Ηνωμένων Βασιλείου, τα λοιπά κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολούνται σε ομάδες ε, χωρών που δεν συμπίπτουν όμως ε, με τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν και γι' αυτό θεωρούμε ότι με την τωρινή κατάσταση περιορίζεται η ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συντονίσει τις θέσεις και να λειτουργήσει από κοινού. Οπότε θεωρούμε ότι χρειάζεται τροποποίηση τη δομή του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να απηχούνται καλύτερα ε, και η διεθνή πραγματικότητα και η διεθνή θέση τη Ένωση. Προτείνουμε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιζητήσει ε, καθεστώς μόνιμου παρατηρητή στο εκτελεστικό συμβούλιο του Διεθνούς Ομισματικού Τμήματο και της Παγκόσμιας Τράπεζας ε, και να εκπροσωπείται οπωσδήποτε στην Παγκόσμια Τράπεζα όταν είναι θέματα ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συζητούνται. Ε, χρειαζόμαστε ένα πρόεδρο για τις, ευρωπαϊκές, ε, ε, για τις χώρες που ανήκουν στη ζώνη ευρώ και έναν πρόεδρο που θα μας εκπροσωπεί στο εκτελεστικό συμβούλιο για τις χώρες που δεν ανήκουν στη ζώνη ευρώ. Έχουν γίνει συζητήσεις στο παρελθόν για το θέμα αυτό δεν έχουμε καταλήξει όμως σε μία λύση. Ε, για μία ή δύο ομάδες ε, χωρών ε, θεωρούμε ότι με τη νέα λύση δεν θα μειωθεί η βαρύτητα της ψήφου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση των νέων ποσοστώσεων. Τώρα, για το εκτελεστικό συμβούλιο υπάρχει μία συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι G20 τον Οκτώβρη ε, για δύο έδρες κρατών μελών που δεν θα λειτουργούν βάσει του συστήματος εκπεριτροπής, ε, αλλά πρόκειται για δύο μεγάλες οικονομίες. Ε, είναι καλή απόφαση βέβαια γιατί αποφάσισαν να εκχωρήσουν τις θέσεις τους, τάχθηκαν κατά του βέτο και επίσης προώθησαν περαιτέρω τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμφωνία αυτή προβλέπει ε, ως προς τις ποσοστώσεις ε, και τις ε, έδρες να αρχίσει να είναι πλήρω λειτουργικό το σύστημα μέχρι το 2020 με διάμεσο σταθμό το 2010. Το 2012 θεωρούμε μια καλή ημερομηνία ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να προτείνει η σύσταση Ευρωπαϊκής Εκλογικής Περιφέρειας στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της Παγκόσμιας ε, Τράπεζας και μετά το 2020 μπορεί να επιδιώξει μια ε, ενιαία έδρα για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. για την Παγκόσμια Τράπεζα. Τα πράγματα είναι παρεμφερή, όπως και για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Βασιζόμαστε στα κράτη-μέλη βάσει του συστήματος εκπροσώπησης με εκλογικές ε, περιφέρειες που όμως ε, δεν οδηγεί σε ικανοποιητική εκπροσώπηση των κρατών μέλων της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Συχνά ομαδοποιούνται κράτη-μέλη με άλλε χώρε που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκπροσωπούνται όλε αυτέ οι χώρε μαζί στο εκτελεστικό συμβούλιο. Άρα δεν μπορεί να υπάρχει ενιαία φωνή, ενιαία εκπροσώπηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ όμω τα πράγματα περιπλέκονται, διότι οι πολιτικέ ε, δεν είναι αμυγό και κοινοτική αρμοδιότητα, είναι θέματα μεικτή αρμοδιότητα. Η Παγκόσμια Τράπεζα δεν έχει όμως αρμοδιότητα για την νομισματική πολιτική, άρα δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα. Θα προτείναμε λοιπόν στην περίπτωση της Παγκόσμιας Τράπεζας το εξή, η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδιώξει μία ενιαία θέση, έδρα διευθυντού στο εκτελεστικό συμβούλιο που θα συμμετάσχει στο μεταρρυθμιστικό ε, πρόγραμμα τη ε, τράπεζα και στην προσχώρηση νέων χωρών, επιδιώκοντα την κατάργηση του βέτο για τη ΣΥΠΑ ε, στο εκτελεστικό συμβούλιο τη Παγκόσμια Τράπεζα. Την ίδια μεταρρύθμιση μπορούμε να εφαρμόσουμε στις πολυμερείς περιφερειακές τράπεζες όπως αυτή της Αφρικής, της Αμερικής, όλες τις περιφερειακές αναπτυξιακές τράπεζες. Τώρα, σε σχέση με τη σύνθεση G20 και τη θέση εκεί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τέσσερα κράτη-μέλη ανήκουν στο G20, ε, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και προσκαλείται μονίμως και η Ισπανία εκπροσωπείται τριπλά δηλαδή η Ένωση σε εθνικό και σε υπερεθνικό επίπεδο. Σε δύο περιπτώσεις ήταν, συμμετείχε η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Σύνοδο Κορυφής G20. Με δύο τρόπους τουλάχιστον μπορούμε να βελτιώσουμε τη θέση της Ένωσης. Πρώτον, οι εκπρόσωποι δεν δηλαδή πρέπει να γίνουν από δύο ένας ε, στις συνόδους του G20. Πρέπει να αποφασίσουμε ποιος από τους δύο πρόεδρους του Συμβουλίου, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα παρευρίσκονται και επίσης θα πρέπει οι πέντε ευρωπαϊκές χώρες ε, και ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα είναι στη Σύνοδο Κορυφής G20 πρέπει να συντονίζουν τι θέσει του τέλο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιδιώξει καλύτερη σχέση, καλύτερο σύνδεσμο μεταξύ του G20 και των Ηνωμένων Εθνών, ε, ούτω ώστε να έχουμε την ομοποίηση των Ηνωμένων Εθνών και στο G20 και προτείνουμε το εξή. Η G20 να είναι ad hoc, ε, ένα ad hoc ε, διυπουργικό εργαλείο που θα συνεργάζεται με το ECOSOC για την εκπόνηση οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών ή Ο πρόεδρο ζητά από τον ομιλητή να μιλά πιο αργά. Ναι, αλλά ολοκληρώνω τώρα, πρόεδρε. Η δεύτερη λιγότερο φιλόδοξη λύση, η βραχυπρόθεσμη λύση, είναι οι δύο οργανώσεις, η σύνθεση G20 και τα Ηνωμένα Έθνη εργάζονται χωριστά και όλη η πλήρη νομιμοποίηση των Ηνωμένων Εθνών να μην μετακυλιστεί στο G20, αλλά ε, οι τελικές αποφάσεις G20 και ΠΟΣΟΚ ε, να εξετάζονται από τα Ηνωμένα Έθνη, να λειτουργούν ως συμβουλευτικοί οργανισμοί δηλαδή, ε, το G20 και το ΕΚΟΣΟΚ. Ε, Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια την κυρία Μουνιέθ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχει διαφύγει από κανένα και κυρίω στην Επιτροπή μας ότι χρειάζεται παγκόσμια διακυβέρνηση για κοινά προβλήματα και σήμερα αυτή χωλαίνει. Υπάρχουν διεθνείς οργανισμοί και θεσμοί που λειτουργούν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, αλλά έχουν πολλαπλασιαστεί τώρα τα θέματα και η περιπλοκότητα τους διεθνώς και μάλιστα ε, με ηλικιώδεις ρυθμούς οι διεθνείς οργανισμοί και τα κράτη βρίσκονται στα όρια της δυνατότητας διαχείρισης αυτών των καταστάσεων. Κινδυνεύουν ορισμένα θεσμικά όργανα, ορισμένοι θεσμοί και οργανισμοί και έχουμε όλο και περισσότερα κλαμπ, λέσχες, επιμέρους ad hoc ε, συνενώσεις κρατών που δεν έχουν πάντα ούτε συνέχεια, ούτε συνοχή, ούτε ε, δημοκρατική νομιμότητα, ούτε υποκαθιστούν τους ε, διεθνείς οργανισμούς. Και επειδή είναι πολύ πολύ πλέον στον κόσμο, χρειάζεται παγκόσμια διακυβέρνηση με στρατηγικό σχέδιο που σήμερα λείπει. Οι παράγοντες κλειδιά έχουν και δυσκολίες με τα ίδια τα εσωτερικά τους ε, σχήματα, όργανα και δομές και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν επειδή υπάρχει δυσκολία διαχείρισης κατάστασης και η συνθήκη της φιλοδοξεί ε, να κάνει παγκόσμιο πρωταγωνιστή και πάλι ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε μια νέα εξωτερική αρχιτεκτονική. Όλα αυτά ε, συνεισφέρουν έτσι ώστε η έκθεση αυτή και τελικά η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το πώς βλέπει το ρόλο του και της Ένωσης διεθνώς είναι πάρα πολύ επίκαιρη και σημαντική συζήτηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, και δεν θα επιμείνω, έχει ένα σχετικό ειδικό βάρος στον κόσμο παντού και ε, στα εμπορικά θέματα και στο ΕΠ και ε, ως στρατιωτική δύναμη, ως βασικός δωρητής στην αναπτυξιακή βοήθεια, ως ε, συνεισφέρουσα στον προϋπολογισμό του ΟΗΕ, με πολλά προγράμματα, με πολλές αποστολές και επιπλέον έχουμε και τη συνθήκη της Λισαβόνας που ε, δίνει μια νέα διάσταση στην εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή όμως η φιλοδοξία της συνθήκης προσκρούει ε, στη δυσκολία και στις αμφισημίες της ίδιας της συνθήκης. Το σύστημα ε, εκχώρησης αρμοδιοτήτων και η θεσμική πολυπλοκότητα, ο λαβύρινθος αυτός, ιδιαίτερα στην εκπροσώπηση την εξωτερική, είναι πρόβλημα. η διεθνής ε, πρακτική και τα τεκτενόμενα στρέφονται ακόμα γύρω από κράτη ε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κράτος. Γι' αυτό ε, προκύπτει μια επιπλέον δυσκολία και χρειάζεται και μεταρρύθμιση της διεθνούς αρχιτεκτονικής για να δούμε πώς θα ενταχθεί ως δομικό συστατικό της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία, έξω και η εκθεσή μου δεν μπορούσε να είναι γραμμική. Αλλά ε, με διαφορετικό τρόπο αντιμετωπίζει τους διάφορους ε, διεθνείς οργανισμούς. Στο σχέδιο αυτό λοιπόν ε, εξετάζω τα προαπαιτούμενα για να δράει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως πρωταγωνιστής παγκοσμίω μετά την Ευρωπαϊκή Συνθήκη της Λισαβόνας. Είναι έξι τα μεγάλα κεφάλαια και χωρίζω και σε υποπαραγράφους. Επιλέγω μια σειρά πολυμερών οργανισμών που ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να έχει μεγαλύτερη παρουσία. Κάνουμε μια σειρά γενικές ε, συστάσεις αλλά και ειδικέ προς τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση στη διεθνή ε, κονίστρα. Ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης λοιπόν ε, στους διεθνείς οργανισμούς και ιδιαίτερα αναφορά στη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να, πώς να, το πω, να αντικατοπτρίζει την παγκόσμια συνεργασία, να είναι και ηγητική στην κοινή δράση για τη ε, διακυβέρνηση και για το χειρισμό για την αντιμετώπιση των παγκοσμίων προκλήσεων. Γίνεται λόγος για τη μεταρρύθμιση των διεθνών αυτών οργανισμών επίσης και πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να επωφεληθεί από αυτές για να ε, ενισχύσει και το δικό της ρόλο και των οργανισμών με στρατηγική εστίαση και κριτήρια ε, συνεκτικά και συνεπής στην εξωτερική εκπροσώπηση με μόνιμη αναθεώρηση των σημερινών ε, συνεννοήσεων και συμφωνιών για την εκπροσώπηση Ευρωπαϊκής Ένωσης. για να αναβαθμιστεί παντού κατά μία βαθμίδα, κατά μία κλίμακα η Ευρωπαϊκή Ένωση και να ενισχυθεί η διεθνής διπλωματία, συλλογική διπλωματία της Ένωσης με τα κράτη-μέλη. Αυτό υπάρχει και στις αποκλειστικές αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως είπαν και εκπρόσωποι εμπειρογνώμονες που έκαναν τη μελέτη, στις αποκλειστικές αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει μία εκπροσώπηση ενιαία, όπως γίνεται στον ΠΟΕ ή στο ΦΑΟ. Ένα αντιπαράδειγμα σε αυτό είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη ε, διάσκεψη για την κλιματική αλλαγή, όπου ε, είναι συντρέχουσες αρμοδιότητες αλλά και αποκλειστικές αρμοδιότητες, αλλά δεν μιλάμε με μία φωνή, ε, έχουμε παραφωνία και πολυφωνία. Στις συντρέχουσες αρμοδιότητες επίσης θα πρέπει να έχει ε, μία έδρα η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση και από μία ε, τα κράτη-μέλη. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών. Καλούμε προς μία ενίσχυση της θεσμικής ισορροπίας, όπως ακούστηκε, ουσιαστική συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση Ο κύριος Φερνάντο Γκυμαράες θα μιλήσει νομίζω, είναι παρόν. Ε, στη Γενική Συνέλευση λοιπόν των Ηνωμένων Εθνών γίνονται ενέργειες για να εγκριθεί ένα ψήφισμα προς την κατεύθυνση αυτή για ουσιαστική πραγματική συμμετοχή διαφορετική από αυτή που είχαμε μέχρι τώρα. Στο Συμβούλιο Ασφαλείας στόχος είναι η μεταρρύθμιση του Ήδη με τα τελευταία γεγονότα, αλλά και τα πιο πρόσφατα, αλλά και τα τελευταία χρόνια έχει φανεί ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν ανταποκρίνεται στις σημερινές απαιτήσει της παγκόσμιας κοινότητας. Και αυτό που μας ενδιαφέρει να έχουμε συμμετοχή και στο Συμβούλιο Ασφαλείας ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό μάλλον είναι ευσεβής πόθος και πολύ μακράς πνοής. Ε, να υπάρχει όμως συντονισμός και διαβουλεύσεις των κρατών μελών της Ένωσης που είναι μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ε, το τρίτο κεφάλαιο αφορά τους διεθνείς οικονομικούς ε, οργανισμούς. Ε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όπου εκπροσώπησε Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τελείως αναποτελεσματική και περιορίζει τη δυνατότητα επιρροής που έχει η Ευρώπη. Παρόλο που έχει και ε, αποκλειστικές αρμοδιότητες σε νομισματικά θέματα, οπότε πρέπει να έχει και μια ε, έδρα στο εκτελεστικό συμβούλιο του Δούνου του. Για την Παγκόσμια Τράπεζα τώρα. Είναι πολύ σημαντικό ε, το καθεστώς που έχουμε παρατηρητού στο Διοικητικό Συμβούλιο και επίσης καλό θα ήταν τα κράτη-μέλη να είναι όλα ενωμένα σε μια ευρωπαϊκή περιφέρεια, constituency. Για τον ΟΑΣΕ τώρα ζητούμε καθεστώς παρατηρητού και στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, στο Συμβούλιο Βορειοατλαντικού Συμφωνού για να ε, προσαρμοστούμε στο πνεύμα της Σύνθεξης Λισαβόνα που ζητάει κοινή πολιτική άμυνας και ε, συντονισμό με τον ΝΑΤΟ. Σε ό,τι αφορά το ΟΑΣΕ η ύπατη εκπρόσωπο θα πρέπει να είναι παρατηρήτρια στον ΟΑΣΕ εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ε, ε, οι πολυμερείς οργανισμοί είναι περίπλοκοι όπως και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Γίνονται όλες οι διαδικασίες με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες νομικές προσαρμογές έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης να μπορεί να κυρώνει και να κυρώσει συμφάσεις ε, προκειμένου την ΕΣΔΑ την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και ε, ξέρουμε ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ε, ιδιαίτερο στο χαρακτήρα του για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα λέει και η συνθήκη αυτά. Και άλλος ε, πολυμερής οργανισμός, σας είπα, είναι ο ΩΣΑ και η Ευρώπη να μην είναι μόνο παρατηρητής αλλά πλήρες μέλος. Και πάλι είναι αποκλειστικές αρμοδιότητες και συντρέχουσες αρμοδιότητες που είναι στον όσα. Έκτον, και άλλο περίπλοκο θέμα και πιο ασταθές. Είναι η διπλωματία των συνόδων κορυφής, το G20 και το G8. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει κανονικά να συμμετέχει σε αυτές τις διαδικασίες και πλήρως να εκπροσωπείται αλλού σε συνεδριάσεις ε, του G7 των Υπουργών Οικονομίας. Και το G20 επίσης ε, κερδίζει όλο και περισσότερο σε σημασία και σε επιρροή. Γι' αυτό θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμμετέχουν ως Ευρωπαϊκή Ένωση σε υπουργικό επίπεδο στις υπουργικές ε, συνόδους κορυφής του G20. Αυτά είναι τα έξι κεφάλαια που σας είπα, έξι ενότητες τις οποίες επικεντρώνεται το σχέδιο εκθεσής μου που βεβαίως ε, είναι στη διάθεσή σας και για τροπολογίες και για τις δικές μου τροπολογίες και απομένουν πολλά στοιχεία να διευκρινιστούν, να συγκεκριμενοποιηθούν, να δοθούν νέες ιδέες. Θέλω να ευχαριστήσω, όπως περιπτώσει, το Ίδρυμα Αλτερνατίβα εναλλακτικέ για τη μελέτη που εκπώνησε και νομίζω ότι σας έχει διανεμηθεί. Είναι πάρα πολύ σοβαρή έκθεση, πάρα πολύ αντικειμενική και αυστηρή με ε, νέες ιδέες χρήσιμες για να μπορέσει το Κοινοβούλιο να λάβει θέση σε αυτό το περίπλοκο θέμα που για πρώτη φορά μας απασχολεί και σε μια στιγμή που είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Και θέλω να ευχαριστήσω και τον Πίτερ Βάσκετ και τον, ε, τη γραμματεία της έκθεσής μας για τη συστηματικοποίηση και για τις συνέργειες που έφερε σε αυτή την έκθεση πολιτικά ασχολούμαι με αυτό το θέμα και από τη γραμματεία για τη ε, Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και θα προσπαθήσω ο συντονισμό που καμιά φορά λείπει μεταξύ κρατών μελών και θεσμικών οργάνων να επιτευχθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή μα μεταξύ των διαφόρων ε, ε, στοιχείων που μας απασχολούν ενός με τους διάφορους πυλώνες. Θα ήθελα να απευθυνθώ και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ασχολούνται με αυτά τα θέματα τη πολυμερούς συνεργασία. μας βοήθησαν πάρα πολύ για να έχουμε μια συνολική θεώρηση ε, του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους διάφορους οργανισμούς και επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους βοηθούς μου και τους συνεργάτες μου που είχαν λίγο χρόνο στη διάθεσή τους αλλά εργάστηκαν θαυμάσια για να μπορέσουμε να καταθέσουμε σχέδιο έκθεσης ε, πιο σύντομο από το αρχικό γιατί έχουμε τώρα κάποιες υποχρεώσεις, κάποιους περιορισμούς χρόνου και χώρου ε, για τη μετάφραση. Μας επιβάλλει ε, ορισμένο αριθμό χαρακτήρων σε μια ε, έκθεση η διοίκηση. Εγώ θα την ήθελα εκτενέστερη, τι να κάνουμε. Ελπίζω να τη βελτιώσουμε μέσω των τροπολογιών. Και με τους σκιώδεις ηγητές ελπίζω να καταλήξουμε σε συμβαστικές τροπολογίες, να κάνουμε την έκθεση αυτή είναι ενετική, διότι νομίζω ότι είναι θέμα θεσμικό. Αυτό που θα πρέπει να βγει από το Κοινοβούλιο είναι μια θέση του θεσμικού οργάνου. Και είναι σημαντικό και το περιεχόμενο και η ουσία και θα συζητηθεί στην Ολομέλεια με παρουσία της κυρίας Άστον και στην ευρύτερη συζήτηση για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμμετοχή της στα διεθνή τεκτενόμενα. Είναι σημαντικό ε, η μεγάλη συζήτηση για την εξωτερική πολιτική να γίνει ουσιαστική και η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να ε, διαδραματίζει το ρόλο που της αρμόζει και της αναλογεί διεθνώς. Ευχαριστώ πολύ. Euh, Σα ευχαριστούμε κυρία Μουνής. Ε, θα δώσω το λόγο τώρα στους ομιλητές που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο. Σας παρακαλώ να μην υπερβαίνετε τα δύο λεπτά κατά αγόρευση. Είναι πολύ φορτωμένη μέρη σε διάταξη. Η κυρία Χάουτα, από την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, δεν θα χρειαστώ πάνω από δύο λεπτά. Κυρία Μούνη, ε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, μας παρουσιάσετε μια, ένα θαυμάσιο σχέδιο έκθεση και αυτό που λέτε να έρθει, είπατε, εκπρόσωπο οποίος ε, με μια, ένα λευκό έγγραφο για τις ε, πολυμερείς σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η πρόταση είναι πάρα πολύ καλή τη στιγμή που εφαρμόζεται η συνθήκη της Λισαβόνας και η υπηρεσία εξωτερικής δράσης ε, έχει ορίσει τις προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία λοιπόν από αυτές πράγματι είναι να ενισχυθεί η πολυμέρεια. Αυτή είναι η στρατηγική ασφαλείας από το 2003. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να εξετάσουμε και το θέμα της της ε, νομιμότητας με την ευρύτερη έννοια, να το συνδυάσουμε με τον εκδημοκρατισμό της παγκόσμιας διακυβέρνησης και πώς μπορεί να στηρίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή την έννοια. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό σχετίζεται άμεσα ε, με την έκθεση του ε, κυρίου Λάμπστορφ, την οποία και θα ακούσουμε σήμερα αργότερα. Ε, νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ε, συμμετοχή και έλεγχος των δραστηριοτήτων, ίσως με την ενίσχυση της Γενικής Συνέλευσης. Εξάλλου, όσον αφορά την νομιμότητα ε, της λήψης αποφάσεων ε, για την πολυμέρεια, ακούσαμε θαυμάσιες προτάσεις για το πώς οι νέε, ε, το G8 και το G9 μπορούν να εκπροσωπηθούν καλύτερα ε, στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών. Εδώ λοιπόν ε, βλέπουμε τον ενισχυμένο ρόλο των αδειόμενων δυνάμεων. Πράγματι θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερο, ισχυρότερο λέγιν στους διεθνείς οργανισμούς. Δεν ξέρω αν μπορούμε να ενισχύσουμε την περίφημη ερεσιμότητα και θα ήθελα να αναφέρω και το θέμα της εξορρόπησης των συμφερόντων και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να ε, αντισταθμίσουμε τα εμπορικά συμφέροντα με άλλα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον και άλλα. Εδώ λοιπόν πρόσφατα το Κοινοβούλιο κατέθεσε μια θαυμάσια έκθεση που πρέπει να έχουμε κατά νου. Ε, πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσουμε τους αναδυόμενους εμπορικούς μηχανισμούς ε, με πιο καινοτόμο τρόπο. Ας μην ξεχνάμε το Google αναφέρθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, σχετικά με το ότι η ε, λογοκρισία του διαδικτύου ε, στο, στην Κίνα μπορεί να αποτελεί και παραβίαση των διατάξεων του ΠΟΕ. Εγώ λοιπόν νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι πολύ πιο ανοιχτή, με μεγαλύτερη κατανόηση απέναντι το Συμβούλιο τη Ευρώπη, τη στιγμή μάλιστα που η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνεται να ε, συμμετάσχει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δεν είχα και άλλη να πω, νομίζω ότι τέλειωσε ο χρόνος μου. Σήμερα Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος ε, Λάμπστορφ τώρα, πρόεδρος ομάδας εργασίας για τις σχέσεις Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και Οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών. Ευχαριστούμε πολύ για την έκθεση της κυρίας Μουνής που τη βρίσκω πάρα πολύ καλή και θέλω να πω ότι εδώ πρόκειται για μια έκθεση η οποία κατά την άποψή μου ε, βασίζεται σε μια μελέτη την οποία έτσι ξεφύλλεις απλώς για να μιλικρινείς που κάνει όμως θαυμάσια εντύπωση. Ε, το θέμα τίθεται τελείως διαφορετικά ε, όπως πραγματικά ισχύει. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι εδώ έχουμε μια διαφοροποιημένη προσέγγιση. Δηλαδή δεν μπορούμε να εμφανιστούμε με τον ίδιο τρόπο σε όλους αυτούς τους ε, διεθνείς οργανισμούς και αυτό αναφέρεται πάρα πολύ καλά στην έκθεση. Εγώ λοιπόν νομίζω ότι η καθυστερημένη αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολύ συχνά καθυστερημένη αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους οργανισμούς είναι ένα πρόβλημα. Και στα αγγλικά πολλές φορές λέμε ε, πράγματι υπερεκπροσωπούμεθα αλλά υπολειτουργούμε. Όντως, ε, πολλές φορές Δυστυχώ, ε, επειδή θέλουμε να εμφανιστούμε παντού, αυτό που κάνουμε είναι απλά να περιζόμαστε σε δραστηριότητε συντονισμού. Και θέλω να πω τα εξή. Όσον αφορά την κατεύθυνση, πράγματι τη συμμερίζουμε. Πολύ καλή η ανάλυση στη μελέτη. Ε, εκείνο που μπορούμε να κάνουμε, ίσω να καταστήσουμε την έκθεση περισσότερο πολιτική. Γιατί όπω είπε και η κυρία Χάουταλα, έχει φτάσει πια η κατάλληλη χρονική στιγμή. Έχουμε αυτή τη στιγμή βέβαια μια κρίση, γι' αυτό και η συζήτηση αφορά περισσότερο ε, τους ε, αφεκιονάντους αυτούς που είναι εξοικειωμένοι με τα θέματα. Όμως εδώ υπάρχει και ένα πολιτικό μήνυμα ότι πρέπει να προχωρήσουμε. Άλμα πρέπει να κάνουμε, σαφέστεροι να είμαστε στα αιτήματά μας και προς τα κράτη-μέλη και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, κυρίως όσον αφορά τον απολογισμό και την υποβολή συστάσεων. Αυτό λοιπόν πρέπει να είναι το μήνυμα το οποίο πρέπει να βγει και από τη συνάντησή μας. Προτείνω πιο συγκεκριμένα τα εξή να διαγραφεί το εδάφιο Α, γιατί θεωρώ ότι το Β είναι πάρα πολύ καλό. Το Α μας δίνει έτσι μια ακαδημαϊκή ιδέα για τις διάφορες διαδικασίες ε, της ε, παγκοσμιοποίησης και τις συστημικές αποτυχίες αυτών των προσεγγίσεων. Εγώ θεωρώ ότι η παγκοσμιοποίηση είναι περισσότερο μια ακαδημαϊκή κουβέντα. Όμως το εδάφη ήταν μια θαυμάσια διατύπωση που μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για ε, είσοδο στο θέμα, για προήμιο στο θέμα. Κατόπιν, δεν ξέρω κατά πόσο πράγματι έχει λάβει η χώρα η μεταρρύθμιση στην Παγκόσμια Τράπεζα στο Διεθνές Δομινικό Έχει λάβει χώρα αυτή η τροποποίηση ξέρω όμως για την Παγκόσμια Τράπεζα. Κατά τα άλλα, ίσως θα βοηθούσε να ε, επισημάνουμε ένα πολύ καλό παράδειγμα όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται θαυμάσια μέσα στην πολυμέρεια. Είναι η ε, επιχείρηση Αταλάντα όπου είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία με το ΝΑΤΟ. Αυτές ήταν οι πρώτες παρατηρήσεις. Θα καταθέσουμε κάποιες ε, τροπολογίες, αλλά έχει σημασία η κατευθυντήρια, η κατεύθυνση που αναλαμβάνει που ακολουθεί, με συγχωρείτε, η έκθεση και αυτή κατά την άποψή μου είναι πάρα πολύ καλή. Ευχαριστούμε κύριο Σκούκεν τώρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να είμαι σύντομος. Το αντικείμενο της έκθεσης είναι τέτοιο ώστε δεν υπάρχουν αντικρούμενα σημεία. Όλοι θέλουμε να ενισχύσουμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωση στη διεθνή σκηνή. Θέλουμε να έχει ηγετικό ρόλο η Ένωση. Δεδομένου των τραγικών εξελίξεων στη διεθνή πραγματικότητα που βιώνουμε σχάτω, είναι λογικό αν θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ε, σε, με ισότιμους όρους να μάλλον να έχει την ίδια θέση όπως η Ινδία, η Βραζιλία, η Κίνα, την ίδια θέση με άλλους παγκόσμιους παίκτες δηλαδή εκ των έσω πρέπει να ενισχύσουμε τη θέση μας και να αναβαθμίσουμε τη θέση μας σε διάφορους ε, διεθνούς ε, οργανισμούς. Η έκθεση της κυρίας Μούνης ε, είναι μια καλή βάση, ένα καλό έρισμα για τις μελλοντικέ μας συζητήσεις. Συμφωνώ και με τους συναδέλφους από την Ισπανία. Δεν είναι ακαδημαϊκή η θέση τους, δεν είναι θεωρητική, αλλά τουλάχιστον κάνουν συγκεκριμένες εισηγήσεις. Και αυτό είναι το γενικότερο μου σχόλιο για το ψήφισμα. Δηλαδή, έχουμε πάρα, πολύ, πάρα πολύ ωραίες ιδέες, ίσως και υπερβολικά πολλές ιδέες. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είναι ακαδημαϊκού χαρακτήρα το έγγραφο, πρέπει να είναι ρεαλιστικό το σχέδιό μας. Να εκπονούμε μια πολύ ε, ουσιαστική πολιτική, να βρούμε τις λύσεις για να υλοποιήσουμε τους στόχους μας. Δηλαδή τέτοιου είδους ψηφίσματα είναι τόσα, τόσο πολύ άριθμα αυτά τα ψηφίσματα και δεν είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε απτά αποτελέσματα ώστε να βελτιώσουμε την κατάσταση μέσω του ψηφίσματος. Σας ευχαριστούμε, κύριος Presidente. Eh, ehm, Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Συγήτρια για την έκθεσή της. Εγώ θα ήθελα να τοποθετηθώ έτσι κάπως ε, γενικότερα, κυρίως ε, διότι πιστεύω ότι η συνθήκη της ε, Λισαβόνας ε, έχει περισσότερο μια ε, προσέγγιση διακυβερνητική. Η αλήθεια είναι ότι η παγκοσμιοποίηση οδήγησε στο να χάσουμε σημαντικά στοιχεία της εδαφικής της κυριαρχίας, εθνικής κυριαρχίας. Κυρίως αυτό αφορά στα κράτη-μέλη. Το θέμα είναι βέβαια ότι ε, δεν ξέρουμε κατά πόσον ε, πράγματι πρέπει η εθνική κυριαρχία να είναι αντικείμενο αντιμετώπισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ναι, να εκχωρηθεί ε, κυριαρχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως κάποια στοιχεία αυτής χάνονται και ο μόνος τρόπος για να τα ανακτήσουμε είναι να την διαχειριζόμαστε με δική μας συγκατάθεση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να ε, δραστηριοποιηθούμε απλά και μόνο επειδή η παγκοσμιοποίηση είναι κάτι το σκληρό ε, και συμμετέχει κανείς σε αυτή την παγκοσμιοποίηση με μέσα και εργαλεία τα οποία συγκρίνονται με αυτά που διαθέτουν οι άλλες ε, μεγάλες χώρες. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό πρέπει κανείς να το έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του ε, και να το λαμβάνει υπόψη του. Το δεύτερο το οποίο θέλω να επισημάνω είναι ο εκδημοκρατισμός. Εκδημοκρατισμός ε, των διεθνών οργανισμών ε, και αυτό πρέπει να το επιδιώξουμε με κάθε δυνατό τρόπο. Ε, όχι μόνο τον εκδημοκρατισμό, αλλά αν θέλετε και τον εξορθολογισμό. Γιατί εγώ προσωπικά πιστεύω ότι όλοι οι ε, θεσμοί του Bretton Woods, δηλαδή η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα πρέπει να ενταχθούν στο ίδιο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, στους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών και επίσης και, στον, και ακόμα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου και αυτός πρέπει να ενταχθεί σε αυτό το σύστημα. Ε, γιατί θα πρέπει βεβαίως και να δίνονται κίνητρα αλλά και να επιβάλλονται και πρόστιμα, κυρώσεις. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν μέσα από το σύστημα, το διεθνές σύστημα. Ως εκ τούτου θεωρώ ότι αυτή πρέπει να είναι η κατεύθυνση την οποία πρέπει να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και με τον τρόπο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει πράγματι να συμμετέχει περισσότερο στον εκδημοκρατισμό αλλά και στον εξορθολογισμό των διεθνών οργανισμών έτσι ώστε πράγματι να σημειωθεί πρόοδος στο θέμα της δικαιοσύνης και της ειρήνης. Σας ευχαριστούμε κυρία Γκόμες τώρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ τη Μαρία Μουνίσε για το εξαιρετικό ψήφισμα που μας υποβάλλει. είναι πλήρες, εντοπίζει τα προβλήματα και προτείνει λύσεις. Η Μαρία προσπάθησε να προτείνει μετριοπαθείς λύσεις ώστε να συλλέξει και τη συνένεση των μελών. Ο ρόλος του Κοινοβουλίου μας, ε, ή μάλλον να θέσω αλλιώς. Πρέπει να δείξουμε μεγαλύτερο θάρρος ε, στο Κοινοβούλιο για να εντοπίσουμε τα προβλήματα και για να προτείνουμε αποτελεσματικέ αποτελεσματικές λύσεις εξηδίας εμπειρίας. Ε, θα έλεγα ότι η μεταρρύθμιση του κογουαστορικού κανονισμού του Συμβουλίου Ασφαλείας έχει κέρια σημασία. Τώρα με τη συνθήκη της Λισαβόνας και τις προβλέψεις και τους στόχους που συνεπάγεται για την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε τη διαφορά. Αν είμαστε πιο θαραλοί, αν πιέσουμε για την τροποποίηση του Συμβουλίου Ασφαλείας, μπορούμε να ενεργοποιήσουμε την διαδικασία, αν συμφωνήσουμε μεταξύ ημών, για τον τρόπο με τον οποίο θα εκπροσωπούμαστε στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Άρα Δεν πρόκειται για μια επανάληψη των θέσεων μα ένα διευρυμένο δηλαδή συμβούλιο να έχει έδρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω έλεγε η Μαρία. Ναι, σημαντικό και αυτό, αλλά είναι ο ελάχιστος κοινό παρονομαστής. Ε, περισσότερα θα έπρεπε να επιδιώκουμε. Αν δεν έχουμε εμεί το όραμα, αν δεν αναλάβουμε εμεί ηγετικό ρόλο στο Κοινοβούλιο εννοώ, ποτέ δεν πρόκειται να προκύψει αυτό από τα κράτη-μέλη. Γιατί βρίσκονται και σε απόγνωση τώρα, πώς να το πω αλλιώς. Πρέπει να είναι πιο θαραλέο το κοινοβούλιο, να συζητήσει τη διεύρυνση, τη δέουσα εκπροσώπηση, τι συνεπάγεται αυτός προ τις ευθύνε μας. Βρίσκω ότι είναι ενδιαφέρον και μάλλον ανησυχητικό που τρεις επιδιώκουν μόνιμη θέση, η Βραζιλία, η Ινδία και η Γερμανία και αυτές οι τρεις δυνάμεις απίσχαν από την ψηφοφορία στο ψήφισμα για την παρέμβαση στη Λιβύη. Δηλαδή τι, θέλουν την ευθύνη, θέλουν μόνιμη έδρα στο Συμβούλιο ασφαλεία και όταν υπάρχει κρίσιμη ψηφοφορία επιλέγουν την αποχή. Πρέπει να ε, είναι πιο καταλητικό, πιο αποφυστικό ο ρόλο μας. Δεν μπορούμε να διαλέγουμε εμεί την αποχή. Για το ΒΕΤΟ, την αρνησή κυρία, δεν μπορεί να υπάρξει ε, πραγματική μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας αν δεν αναθεωρηθούν ε, τα περιβέτο, γιατί ε, παραλύει το Συμβουλίο Ασφαλείας συχνά λόγω του βέτο. Υπάρχουν και άλλα πολύ εύστοχα στοιχεία μέσα στην έκθεση, αλλά θέλω να είμαστε πιο θαραλέοι, πιο τολμηροί στο Κοινοβούλιο και γι' αυτό θα κάνω σχετικές προτάσεις. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Γκέλε. Äh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστώ την κυρία Μινής ε, για την έκθεση που μας ε, παρουσίασε. Εγώ θα ήθελα ε, να εστιάσω την προσοχή μου σε δύο παραγράφους, καταρχήν στα σημεία υπερθυμών 11 και 12. Βεβαίως υποστηρίζω κατηγορηματικά και ανεπιφύλακτα το σημείο 11 ως έχει. Ελπίζω μόνο επιτόπου όσοι λάβουν τις αποφάσεις την επόμενη φορά ε, να μεριμνήσουν καλύτερα. Δηλαδή, όταν θα τεθεί το θέμα του να μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει το λόγο στη Γενική Συνέλευση, ελπίζω τα πράγματα να είναι καλύτερα οργανωμένα. Θέλω να ελπίζω ότι αντλήσαμε διδάγματα από τα λάθη μας ε, όταν ήμασταν στην Κινσάσα, στην συνέλευση των ΑΚΕ ε, η Υπουργό Ασκογιάννα εξήγησε ακριβώς ε, τι θα γίνει και αυτό ήταν απαράδεικτο. Δηλαδή, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μία ημέρα πριν από την ψηφία στην Κογιάννα εμφανίστηκε εκεί και είπε αύριο ε, θα ψηφίσετε προφανώς ως ομάδα ΑΚΕ από κοινού με εμάς. Αυτό έγινε μία μέρα νωρίτερα και είπανε μα με συγχωρείτε εμείς διαφορετικά ε, σχηματίζουμε άποψη. Δεν γίνεται από σήμερα σε αύριο να κάνουμε αυτό που θέλετε και τα πράγματα δεν πήγαν καλά. Ελπίζω λοιπόν ότι τα πράγματα θα αλλάξουν και ελπίζω στο μέλλον να υπάρχει και καλύτερη οργάνωση. Νομίζω λοιπόν ότι στο σημείο 12 θα πρέπει εκεί να είμαστε λίγο περισσότερο φιλόδοξοι. Και όχι μόνο να καλούμε τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ε, συμμετέχουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας να εξηγούν στους άλλους τι ακριβώς συμβαίνει. Εντάξει, καλό και αυτό, όμως ε, πιστεύω ότι από τότε που έχουμε τη συνθήκη της Λισαβόνας και από τότε που θέλουμε ή αποφασίσαμε να έχουμε μια κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, οφείλουμε να έχουμε μια τέτοια προσέγγιση που θα οδηγήσει στο τα κράτη-μέλη τα οποία εκπροσωπούν στο Συμβούλιο Ασφαλείας να εκπροσωπούν την γνώμη όλων. Όπως ακριβώς κατορθώνουμε στο Συμβούλιο Υπουργών να επιτύχουμε κοινέ θέσει ή και σε άλλα συμβούλια με τον ίδιο ακριβώς τρόπο ε, θα πρέπει ε, να γίνεται και το ίδιο ε, στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Να υπάρχει κοινή στάση στις ψηφοφορίες.